Ε, Ημερήσια διάταξη που είναι το μικρό και η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισηγητής κύριος Ντε σας καλώ να λάβετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως για τους υπηρογνώμονες αυτές που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είδαμε στην ομάδα ε, υψηλού επίπεδου είναι ότι είχαμε εκπροσώπους κυρίως από την αυτοκινητοβιομηχανία οι οποίοι συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δεν ακούγεται η φωνή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που υπερασπίζονται το περιβάλλον για τις μη καπαόμικρον αυτές είναι πολύ δύσκολο να ε, μιλήσουν ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές φορές θα πρέπει να πιέσουμε πολύ για εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε υπερεκπροσώπηση των διαφόρων λόμπι σε επίπεδο συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν πως εγώ, επειδή ακριβώς είχα και άτυπες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την προηγούμενη νομοθεσία, πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 καταλήξαμε σε αδιέξοδο. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα πρέπει εμείς να ε, υποδείξουμε σε ποιες περιπτώσεις η, η, σύνθεση δεν ήταν η κατάλληλη, αλλά νομίζω πως σε αυτό θα έπρεπε να το αντιστρέψουμε για γιατί βέβαια στη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μόνο ένας ο υπάλληλος ο οποίος τότε παρακολουθούσε το θέμα αυτό, δηλαδή τη σύσταση και τη σύνθεση αυτών των ομάδων εμπειρογνωμένων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν θα πρέπει να σπρώξουμε το θέμα αυτό κάτω από το ε, χαλί και στη δική μας Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ε, καταλήξαμε πως χρειάζεται μια έκθεση, μια μελέτη η οποία κατέληξε σε αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν, υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας, μια μια ξεκάθαρη έλλειψη ισορροπίας και θα λαμβάνεται υπόψη το θέμα της ε, πρόσβασης στα πρακτικά των διαφόρων συνεδριάσεων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας υποσχέθηκε πως θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά να σας πω πως ποτέ δεν ήρθαν σε επαφή επίσημα μαζί μας. Ή επίσημα μάλιστα μπορώ να σας πω. Γνωρίζουν την ε, θέση μας, ξέρουν πως εμείς θα προετοιμάσουμε και μια σχετική γνωμοδότηση και το το κείμενο το οποίο έχω εγώ, που είναι το κείμενο εργασίας, έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε σχόλια γραπτά. Κάναμε και με τον αντιπρόεδρο κ. Τίμερμανς ε, κάποιες συναντήσεις, είχαμε κάποιες ανεπίσημες επαφές σε θετικό πνεύμα, αλλά δυστυχώς δεν ελήφθησαν όλες τις παρατηρήσεις μας υπόψη και γι' αυτό έχουμε την έκθεση εδώ που χρειάζεται. Ξεκάθαρα κριτήρια για τον ορισμό της πραγματογνωμοσύνης που επιδιώκει να βρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, θα πρέπει ε, όλες οι απόψεις να εκπροσωπούνται στις ομάδες αυτές έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Τρίτον, ένα σύστημα που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και οποιασδήποτε ενστάσει προσφυγές. Τέταρτον, όχι μόνο διπορικά αλλά και οι υπόλοιπε δαπάνες ε, θα πρέπει να πληρώνονται έτσι ώστε να μπορεί και η κοινωνία των πολιτών με εύκολο τρόπο να μετακινείται και να ε, συμμετέχει. Ρόλος των ΜΚΟ μικρών θα πρέπει να ε, στηριχθεί και επίσης ειδική πλειοψηφία Όταν υπάρχει κάποια αντίρρηση για τη δημοσίευση των πρακτικών, θα πρέπει να ξεκάθαρει κανόνες για το πώς θα δημοσιεύεται και με ποιες λεπτομέρειες και επίσης σύγκρουση συμφερόντων και εδώ ξεκάθαροι κανόνες έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποια κύκλοι συμφερόντων που να πιέζουν. Και επίσης ένα όργανο παρακολούθησης έτσι ώστε όλοι αυτοί οι κανόνες να γίνουν σεβαστοί. Αυτά τα συζητήσαμε και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα δει αυτά, θα διαβάσει τη δική μας έκθεση και πριν από την 1η Ιουλίου θα δράσει. Θέλουμε λοιπόν την διαφάνεια την οποία και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανονικά θα έπρεπε να επιδιώξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έλλειψη διαφάνειας και η μη ισορροπημένη σύνθεση πολλών ομάδων εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση αυτών των ομάδων δεδομένου ότι η έλλειψη διαφάνεια έχει αρνητικέ επιπτώσει στην εμπιστοσύνη των πολιτών των κρατών μελών τη ένωση ω προ τα θεσμικά όργανα τη η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματο των ομάδων εμπειρογνωμόνων τη επιτροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τι αρχέ τη διαφάνεια και τη ισορροπημένη σύνθεση. ήδη από την 30 η μαου το 2016 η Επιτροπή είχε θεσπίσει οριζόντιες κανόνες σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να γίνονται δημόσιες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών των ομάδων αυτών και επομένως αυξάνεται η διαφάνεια. Τέλος, το Μητρό των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχει σαν στόχο να αυξηθεί επιπλέον η διαφάνεια στις ομάδες αυτές και να διευκρινίσει τους τρόπους για το πώς πραγματικά θα ενθαρρυνθούν οι υποεκπροσωπούμενες οργανώσεις των κοινωνικών ομάδων για να συμμετάσχουν στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πολύ, četla ony návrhy hledající

Η Επιτροπή όμως δεν προέβη κάποια δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό. Είναι όμως αυτό πάρει πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε για τη σωστή εκπροσώπηση και των κοινωνικών εταίρων. Θα έπρεπε να κάνει κάποια μικρά βήματα η Κομισιόν προς τα εμπρός. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε για πολύ πιο σοβαρά θέματα αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος κυρία Βέσταγκερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, εξωτομοβουλευτές, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντεγιόγκ, και για την έκθεσή του και για το έργο του πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι συμφωνούμε ε, σε σχέση με τους κανόνες και την σπουδαιότητα που έχουν για την ομοποίηση αυτών των συμβουλευτικών ομάδων ε, και των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία χάραξη πολιτικής και έχουμε προβλέψει αυστηρότερους εσωτερικούς κανόνες ώστε να μπορούν αυτές οι ομάδες να φέρνουν σε πέρα στα καθήκοντά τους με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία ακριβώς όπως έχει ζητηθεί. Θα ήθελα να τονίσω ένα μόνο πράγμα που αποτελεί και κάτι στοιχειώδες. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων παρέχουν χρησιμότατες ε, συνεισφορές ε, στο έργο της Κομισιόν σε πολλούς τομείς πολιτικής. Άκρος τεχνικούς ενίοτε ή εξειδικευμένους. Όμως, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επενθυμίσω ότι ό,τι συμβουλές και αν δίνουν αυτές οι ομάδες συμπειρογνωμόνων, ο ρόλος τους είναι αμυγός συμβουλευτικός. Οτιδήποτε συμβουλή λοιπόν μπορεί να παρέχουν, η ευθύνη λήψη οποιασδήποτε απόφαση, οποιοδήποτε μέτρου παραμένει μόνο αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα, αποφασίσαμε ότι οι κανόνες ε, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να ανταποκριθούν ε, περισσότερο στη δέσμευση της Κομισιόν για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Πριν εγκριθεί νέα δέσμη κανόνων, ακούσαμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο διαβουλεύσεων και εταιρική έντονη διεργασία, εγκρίναμε πέρυσι το Μάιο αυτού του νέου κανόνε. Θεωρούμε πω οι νέοι αυτοί κανόνε, που είναι και δεσμευτικοί για όλε τι υπηρεσίε τη Κομισιόν, βελτιώνουν ή θα βελτιώσουν σημαντικά την ισορροπία και τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμών. Θεωρούμε επίσης ότι έτσι ανταποκρινόμαστε θετικά σε πολλές από τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Διαμεσολαβήτριας. Για να σας δώσω λίγα συγκεκριμένα παραδείγματα, οι νέοι κανόνες επανεπιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Κομισιόν για ισορροπημένη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Και θα πρέπει και τα τμήματα τα διάφορα της Κομισιόν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, την πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση Ισορροπημένη εκπροσώπηση δεν σημαίνει μαθηματική ισορροπία, κάτι που βέβαια είναι δύσκολο να οριστεί και να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μαστικά σημαίνει τη μέγιστη δυνατή ισορροπία σε ό,τι αφορά ε, την εμπειρία, τα συμφέροντα, ενδιαφέροντα, γεωγραφική ε, προέλευση, φύλλο κτλ. Επίση, με του νέου κανόνε τονίζουμε ότι έχουμε προωθήσει πολύ περισσότερη διαφάνεια, έχουμε ένα νέο μητρό ε, για τι ομάδε συμπυρογνωμόνων που είναι προσβάσιμο στο κοινό και δίνει πιο ακριβές πληροφορίες ε, παρέχει δε πρόταση στα έγγραφα τα οποία συζητούνται στι ομάδε συμπεριγνωμόνων. κομμησιών, μάλιστα θα δημοσιοποιεί και τους, ε, ε, τις προκηρύξεις διαγωνισμών και θα λέει ποια είναι τα μέλη των ομάδων υπερογνωμόνων που έχουν οριστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τα Και ήταν και ένα μακροχρόνιο έτοιμο του Κοινοβουλίου. Με άλλα λόγια η, επιλογή, διαδικασία επιλογής πλέον είναι εντελώς διαφανής. Και αυτό σίγουρα διευκολύνει και την ισορροπημένη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμών. Δεύτερο, καταγραφή στο Μητρό Διαφάνειας αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τις οργανώσεις εμπλεκομένων φορέων που θα ορίζονται σε μια ομάδα εμπειρογνωμών. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρχει πλήρες διαφάνειας ό,τι αφορά τα συμφέροντα όλων αυτών. Τρίτον, κάθε έγγραφο παράγει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ε, μπαίνει σε αυτό το μητρό, θα αναφέρονται επίσης τα πρακτικά και επίσης οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα μπορούν να αποφασίσουν να συνδυάζουν δημόσια. Τέλος. Έχουμε λάβει πολύ σκληρά μέτρα για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Με τους νέους κανόνες οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να οριστούν μόνο με βάση τυποποιημένων ε, αξιολογήσεων σύγκρουση συμφερόντων, με βάση δήλωση που θα υποβάλουν. Και μόνο αν υπηρεσίε της Κομισιόν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούν να οριστούν με προσωπική ιδιότητα αυτή η εμπειρογνώμηση. Και όλες οι δηλώσεις ε, σύγκρουση συμφερόντων των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα καταχωρίζονται σε αυτό το Μητρό Ομάδων Εμπειρογνωμόνων. Με αυτού λοιπόν τους νέους κανόνες μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε ότι ε, πλέον εκπληρώνεται ο στόχος, ο κοινός στόχος Κομισιόν και Κοινοβουλίου, δηλαδή για μεγαλύτερη διαφάνεια λογοδοσία για τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει τα ναρά αυτούς τους νέους κανόνες ε, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι και εσείς ε, θα ασκήσετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκείτε και θα συνεχίσουμε και εμείς τον διάλογο μαζί σας για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση και για να παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.